La sessione è ripresa. Ξεκινάει η σύνοδος, συνεχίζεται η σύνοδος. Παρακαλώ καθίστε, έχουμε μια μεγάλη μέρα ψηφοφορίες και σήμερα θα προσπαθήσουμε να επιτελέσουμε το καθήκον μας όσο δυνατόν πιο ευχάριστα και γρήγορα. Να χαιρετήσω τον Μαρτίν Σούλτ, απερχόμενο πρόεδρο και να τον ευχαριστήσω για το έργο του σας εύχομαι, όπως έκανα και στη συνάντηση που είχαμε, ό,τι καλύτερο για την πολιτική σας δρομή στη Γερμανία. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την εκλογή των αντιπροεδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχω λάβει τις ακόλουθες υποψηφιότητες.